Possiamo cominciare la Ξεκινάμε λοιπόν. Ξέρετε ότι όπως συνήθως θα μεταδοθεί η συνεδρίαση με το διαδίκτυο. Λοιπόν, έχει ήδη διανεμηθεί η ημερήσια διάταξη συμφωνήσαμε στην έκτακτη συνάντηση της 14ης Μαρτίου η ψηφοφορία για τα πολιτικά κόμματα να γίνει αύριο μετά τις 11 εν Βέβαια θα πρέπει να το συζητήσουμε και οι συντονιστές στο συγκεκριμένο θέμα, αλλά ο κ. Ντάφ έχει στήσει το λόγο. Όπως είπατε, έγινε μια έκτακτη συνάντηση πραγματικά έκτακτη. είναι ότι η έκθεση της κυρίας Γιαννάκου μέχρι τώρα τουλάχιστον δεν έχει οριμάσει επαρκώς για να περάσουμε σε ψηφοφορία. Και θα ήταν σωστό να είμαστε προσεκτικοί. και να περιμένουμε. Πράγματι, λέει ο Πρόεδρος, έχω ήδη πει και εγώ ότι προβλέπεται η ψηφοφορία αύριο, η έκθεση της κυρίας Γιαννάκου, αλλά μιας και έχουν έρθει στην επιφάνεια κάποιες συζητήσεις την τελευταία μας συνάντηση, αύριο το πρωί σε επίπεδο συντονιστών θα αποφασίσουμε αν θα ψηφίσουμε ή όχι. Αύριο το πρωί οι συντονιστές λοιπόν και εσείς ήδη εκφράσατε την άποψή σας, επανέρχεται ο κύριος Ντάφ. θα μπορούσαμε να, να πάρουμε την απόφαση για το αν θα ψηφίσουμε ή όχι αύριο το πρωί, αλλά θα ήταν προτιμότερο και περισσότερο διαφανές η απόφαση αυτή να ληφθεί τώρα. Κοιτάξτε, στην τελευταία μας συνάντηση αποφασίστηκε να ψηφίσουμε. Και γι' αυτό είπα εγώ να περιμένουμε μέχρι αύριο ε, για να συζητήσουμε καλύτερα. Ο Μέσερ Σμιτ. σε επίπεδο σκιωδών την προηγούμενη εβδομάδα και μιας και δεν είναι και μαζί μας η κυρία Γιαννάκου εδώ, συμφωνόμεν με τον κύριο Ντάφο ότι η διαδικασία μέχρι τώρα ήταν χαοτική κάπως και αν δεν συζητήσουμε σήμερα δεν θα μπορέσουμε αύριο να πάρουμε τις αποφάσεις που απαιτείται. Γι' αυτό θα ήθελα να υπάρξει αναβολή της ψηφοφορίας αυτής ε, μέχρι ότου έχουμε περισσότερη ε, συζήτηση, περισσότερο χρόνο για συζήτηση και επικοινωνία. Σάπλιν. Δεν είμαι υπέρ ή κατά. Το μόνο που φοβάμαι είναι ότι είμαστε πραγματικά πάρα πολύ λίγοι. Θα μπορούσε να αμφισβητηθεί η όποια απόφαση να αμφισβητηθει οποια αποφαση παρουμε σε επίπεδο δηλαδή διαφάνειας του τρόπου λειτουργίας μας πρέπει να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Έχνερα, αλλά θέλω να σημειώσω εδώ κάτι. Ενθυμίστε ότι στα πλαίσια της συζήτησης που κάναμε πάνω στο θέμα αυτό στην τελευταία συνάντησή μας, ο λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε να κάνουμε μια έκτακτη συνεδρίαση Μάλιστα στην αρχή είχαμε πει Τετάρτη μεσημέρι και μετά είπαμε την Πέμπτη αλλά η Επιτροπή ήταν κατά. Εν πάση περιπτώσει η κυρία Γιαννάκου το πρωί της Τρίτης δεν μπορούσε να είναι παρούσα. Όταν η απόφαση βγήκε λοιπόν, έτσι ώστε να παραμείνει στην ημερήσια διάταξη συγκεκριμένη έκθεση η Τρίτη το πρωί, η κυρία Γιαννάκου είπε ότι θα άλλαζε τους υποχρεώσεις της έτσι ώστε να μπορέσει να είναι παρούσα. Και καταλαβαίνετε τώρα ότι μιας και η συγγήτρια έχει αλλάξει τις δικές της υποχρεώσεις για να είναι παρούσα, ε, νομίζω ότι θα ήταν προτιμότερο να μπορέσουμε να πάρουμε τις αποφάσεις που χρειάζεται αύριο. Αυτή είναι η άποψή μου, αλλά θα δώσω το λόγο πρώτα στον κύριο Έχνερ. Κύριε Πρόεδρε, δίκιο έχετε όταν λέτε ότι πρέπει να συνδυαστούν εδώ πολλές διαφορετικές απόψεις και συνιστώσεις. Βεβαίως έχουμε λάβει υπόψη μας εδώ το πρόγραμμα και τις δυνατότητες της κυρίας Γιαννάκου που είναι και η συγγήτρια. Θεωρώ όμως ότι πέρα από τα προσωπικά προγράμματα και χρονοδιαγράμματα αυτό που είναι σημαντικό είναι να δούμε αν η Επιτροπή σαν επίσημος θεσμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι σε θέση να αποφασίσει. Πρόκειται για μια απόφαση που πρέπει να προετοιμαστεί σωστά και για το τι θα κάνουμε ακριβώς, ποια σημεία θα γίνουν αποδεκτά, ποια όχι. Θα πρέπει να επεξεργαστούμε σωστά τις συμβαστικές τροπολογίες, έχουν ακουστεί απόψεις και εδώ στην Επιτροπή είδαμε ότι δεν μπορέσαμε να έχουμε μία ουσιαστική συνάντηση με την εισηγήτρια έτσι ώστε να ξεκαθαριστούν αυτά τα επίμαχα σημεία. Χαίρομαι ιδιαίτερα που η κυρία Γιαννάκου θα μπορέσει αύριο να είναι εδώ, αλλά χωρίς την προετοιμασία που χρειάζεται νομίζω ότι δεν είμαστε αυτή τη στιγμή σε θέση να αποφασίσουμε, άρα να ψηφίσουμε. Χαίρομαι ιδιαίτερα που θα είναι αύριο εδώ γιατί τουλάχιστον θα ανταλλάξουμε απόψεις. Ο κύριος Νταφ ζητάει το λόγο. Κοιτάξτε, για να μην χάνουμε χρόνο. Εγώ δεν σας προτείνω να ψηφίσουμε. Εγώ μιλάω για τη διαδικασία. Και εγώ πιστεύω μαζί σας ότι δεν θα ήταν καλό να ψηφίσουμε εφόσον η συζήτηση δεν έχει οριμάσει. να αναβάλουμε λοιπόν, αλλά δεν θα πρέπει νομίζω να αποφασίσουμε τώρα. Η απόφαση μπορεί να ληφθεί αύριο το πρωί. Ε, είμαι κατά λοιπόν του να λάβουμε απόφαση πάνω σε αυτό τώρα. Ας μην αποφασίσουμε τώρα. Νταφ. Κοιτάξτε, οι πολιτικές ομάδες πρέπει να προετοιμαστούν σωστά για μια τόσο περίπλοκη ψηφοφορία. Και δεν έχουμε τον χρόνο για να το κάνουμε. Δεν μπορούμε να προετοιμαστούμε έγκαιρα. Υπάρχουν 400 τροπολογίες οι συμβιβαστικές τροπολογίες δεν είναι πραγματικά συμβιβαστικές, είναι χαοτικές και περίπλοκες και λυπάμαι που η συγγήτρια αναγκάστηκε να αλλάξει και τις ρυθμίσεις για το ταξίδιο της. Νομίζω ότι μπορούμε όμως να έρθουμε σε επαφή της τηλεφωνικά και να της εξηγήσουμε ακριβώς ποια είναι η κατάσταση. Νομίζω ότι η αξιοπιστία και η ακεραιότητα της φήμης μας υπονομεύεται αν προχωρήσουμε πρόσεκτα. Και γι' αυτό κύριε Πρόεδρε θα ήθελα να σας ζητήσω να προασπίσετε την ποιότητα της εργασίας μας. Είμαι υπέρ της αναβολής την Πέμπτη ήρθε στην επιφάνεια ότι υπάρχει μια κάποια αβεβαιότητα θα έλεγα σχετικά με την ουσία και το νόημα σε σχέση με τις λεγόμενες ε, σε εισαγωγικά ρήτρες διακρίσεων. Μας είπε ορισμένα πράγματα στην αρχή και ε, μετά αυτό φάνηκε να μην ισχύει. Εμπασπέτως δεν θέλω να επιμείνω σε αυτό γιατί δεν είναι παρούσα εδώ οπότε δεν θα ήταν σωστό. Κοιτάξτε, ας κλείσουμε. Η άποψή μου, την οποία υποβάλλω στην έγκρισή σας, η πρότασή μου δεν είναι να ψηφίσουμε τώρα, αύριο. Εγώ σας ζητώ να αποφασίσουμε αύριο το πρωί στην ε, συνάντηση των συντονιστών αν θα αναβάλουμε ή όχι την ψηφοφορία. Δεν ξέρω. Εγώ έχω τη γνώμη που έχει και ο κύριος Σέπλινγκ. Δεν είμαι ούτε υπέρ ούτε κατά. Το θέμα είναι σοβαρό, το θέμα είναι περίπλοκο και χρήζει περισσότερης επεξεργασίας. Αλλά γιατί να αποφασίσουμε τώρα και όχι αύριο το πρωί, ο κύριος Μέσσερ Σμιτ. Θα είμαι σύντομος. Ο λόγος για τον οποίο είπα ότι πρέπει να αποφασίσουμε τώρα είναι ότι είμαστε ακριβώς στο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Τώρα θα πρέπει να αποφασίσουμε αν αύριο θα ψηφίσουμε ή όχι. Εγώ δεν λέω ότι αν τυχόν πάρουμε την απόφαση αύριο θα είναι η κατάσταση εντελώς διαφορετική, αλλά θα είναι δύσκολο να μπορέσουμε μέσα σε δύο ώρες, αν ας πούμε αποφασίσουμε να ψηφίσουμε θετικά αύριο, ε, να πάρουμε σωστές αποφάσεις σε σχέση με τις συμβιβαστικές τροπολογίες κτλ. Γι' αυτό λοιπόν εγώ προτείνω να αλλάξουμε το 9 και ίσως αύριο και η κυρία Γιαννάκου να μας δώσει κάποιες εξηγήσει γιατί υπάρχουν πάρα πολλά διφορούμενα στοιχεία στα οποία απαιτείται να έχουμε περισσότερες γνώσεις. Πολύ σύντομα, αν είναι τόσο σαφές και τουλάχιστον ακούγοντας τα μέλη της Επιτροπής αυτό διαπιστώνω ότι είναι θέμα προστασίας της ποιότητας και της αξιοπιστίας της εργασίας μας. Νομίζω ότι ίσως πρέπει να το πούμε στην κυρία Γιαννάκου, γιατί αν κατάλαβα καλά για εκείνη είναι σημαντικό να ξέρει αν θα ταξιδέψει ή αν δεν θα ταξιδέψει. Ίσως λοιπόν πρέπει να της το πούμε ότι μάλλον δεν θέλουμε να ψηφίσουμε αύριο. Una è quella di dire votiamo. Κοιτάξτε, δύο είναι οι λύσει. Είτε θα ψηφίσουμε αμέσω, όχι επί τη ουσία, αλλά όσον αφορά την ε, αφαίρεση αυτού του σημείου σε σχέση με τα κόμματα και τα πολιτικά ιδρύματα και η άλλη λύση είναι να μην αποφασίσουμε σήμερα για αυτό το σημείο αλλά αύριο το πρωί. Ποιοι... Λοιπόν, τώρα πρέπει να αφαιρέσουμε από την ημερησία διάταξη το σημείο 9 ή όχι. Ποιοι είστε υπέρ του να βγει το σημείο από την ημερήσια διάταξη. Σήμερα ή αύριο. Ο κύριος Έφνος νόμιζα ότι είχε πει κάτι άλλο, μπας περιπτώσει. Εγώ ήθελα να αναβληθεί η ψηφοφορία. Αλλά αυτό θα είναι δύσκολο αν είναι παρούσα η εισηγήτρια. Λοιπόν, τώρα, Εγώ θα είχα προτιμήσει να ψηφίσουμε αύριο το πρωί. Ποιοι είναι υπέρ αυτή τη εγώ ο ίδιος. Να πούμε δηλαδή ότι πρέπει να το συζητήσουμε αύριο το πρωί, αν θα αναβάλουμε ή δεν θα αναβάλουμε. Αύριο το πρωί να το συζητήσουμε. Εντάξει, την πλειοψηφία θα δούμε. Ωραία. Πόσους ψήφους έχουμε, πόσες ψήφους έχουμε. Ah, Εγώ απέχω, παρακαλώ να το καταγράψετε, Πρόεδρε. Εντάξει. Λοιπόν, πάντως κέρδισε η άποψη του να αφαιρεθεί το σημείο από την ημερήσια διάταξη και έτσι τελειώσαμε. Άλλο ένα θέμα ήταν από τον Αντιπρόεδρο Λεφτύπ που ήθελε η συζήτηση για την θεσμική, στις θεσμικές θέσεις να ξεκινήσει αύριο στις 10. Αύριο το πρωί οι συντονιστές θα αποφασίσουν νομίζω, όχι εμείς τώρα. Τι λέτε, σύμφωνοι? Ωραία. Όσον αφορά τα σημεία 6 και 9 της ημερήσια διάταξης, που αφορούν την ερμηνεία των άρθρων 156 και 161 του κανονισμού δεν έχει ετοιμαστεί το σχετικό έγγραφο και άρα δεν μπορούμε να το συζητήσουμε. Και αυτό λοιπόν αναβάλλεται για μια άλλη συνεδρίαση. Οπότε τώρα εγκρίνουμε την ημερησία διάταξη με αυτές τις αλλαγές. Ε, no, l'unica cosa riguardo alla questione del rapporto ε, το μόνο για την έκθεση Νομίζω θα πρέπει τουλάχιστον τηλεφωνικά να την ειδοποιήσουμε πως δεν θα γίνει. Αν έρθει έτσι κι αλλιώς, εντάξει, θα το ξανακουβεντιάσουμε. Ανακοινώσει του Πρόεδρου. Οριστικό χρονοδιάγραμμα για τις συνεδριάσεις ε, της Επιτροπής μας για το 2003 υπάρχει στους φακέλους σας επιβεβαιώθηκε η έκτακτη συνεδρίαση της Δευτέρας 14, Οκτωβρίου το απόγευμα. Μια επιπλέον ήταν η συνεδρίαση αυτή. 14 Οκτωβρίου το απόγευμα. Και ως ήθιστε στους φακέλους σας θα δείτε στο σημείο 2 την ενημέρωση που, κάνουν κάνει η γραμματεία μας και που αφορά την κατάσταση επικύρωσης για τα διάφορα κράτη-μέλη και τις ε, συνθήκες αυτές που αφορούν τη διακυβέρνηση και την ε, ένταξη της Κροατίας. Ας περάσουμε στο επόμενο σημείο που είναι η έγκριση των πρακτικών και εδώ νομίζω πως ε, ως ήθιστε η σιωπή σα για τα πρακτικά 17 και 18 Δεκεμβρίου και 21 η και 22 Ιανουαρίου 2013 θα σημαίνει πως εγκρίνονται και μπορούμε να περάσουμε έτσι στο επόμενο σημείο Τη παρουσία της κυρίας Γένσεν, που είναι η συγγήτρια για τον Γενικό Προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης για την περίοδο 2014, τη χρήση 2014. Εμείς ως Επιτροπή δεν έχουμε κάποια αρμοδιότητα που να επηρεάζει εντόνως το προϋπολογισμό, αλλά είναι σωστό να ακούσουμε και εμείς και να πούμε τη γνώμη μας. Γι' αυτό και θα ευχαριστήσω την κυρία Γένσεν που είναι παρούσα και θα της δώσω το λόγο για να μας ενημερώσει. Έπειτα ο συνάδελφος μέσα μετά πει δύο λόγια και μετά όποιος θέλει μπορεί να πάρει το λόγο. Παρακαλώ κυρία Γένσεν. Σας ευχαριστώ πολύ. Και ευχαριστώ που με καλέσατε σήμερα. Επισκέπτομαι όλες τις επιτροπές και βέβαια ορισμένες έχουν περισσότερες γραμμές του προπολογισμού, είναι υπεύθυνε μάλλον για περισσότερες γραμμές από ό,τι άλλες. Ωστόσο πιστεύω πως είναι σημαντικό να υπάρχει αυτός ο διάλογος πριν από τις διαπραγματεύσεις για τον προπολογισμό. Ψηφίσαμε την περασμένη εβδομάδα για τις κατευθυντήριες γραμμές για τον προπολογισμό του 2014 καθώς και για το ψήφισμα για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014 με 2020. Και φυσικά οι κατευθυντήριες γραμμές αντικατοπτρίζουν ότι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση αβεβαιότητας. Δεν έχουμε PDP ακόμα συμφωνημένο, οπότε δεν ξέρουμε τι είδους πλαίσιο, σε τι είδους πλαίσιο κινούμαστε. Δεν έχουμε βάση νομοθετική και γι' αυτό και επικρατεί μεγάλη αβεβαιότητα για το τι θα, κανόνες θα διέπουν τον προπολογισμό του 2014. Και έπειτα στις κατευθύντριες γραμμές υπάρχει και αυτή η επαναλαμβανόμενη συζήτηση που αφορά τις πληρωμές ότι δηλαδή δεν θέλουμε να μπούμε στο 2014 με ένα μεγάλο όγκο απλήρωτων λογαριασμών από το 2012-2013. Θα πρέπει αυτό το πρόβλημα να έχει λυθεί φέτος και ελπίζουμε στο πρώτο ήμιση του έτους. Για τη διαδικασία αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι αύριο θα είναι ο πρώτος τριμερής διάλογος ανάμεσα στο Συμβούλιο, την Ιρλανδική Προεδρία, μια αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου και της Κομισιόν. Και αυτό βασικά έτσι ώστε να ξεδιαλύνουμε πώς θα προχωρήσουν οι συζητήσεις για τον προϋπολογισμό, γιατί θα είναι ενδιαφέρον για την Επιτροπή Ε, ότι φαίνεται πως το Συμβούλιο δεν έχει ανακαλύψει πως υπάρχει συνθήκη της Λισαβόνας. Ε, κάνουν το ίδιο που έκαναν και με το παλιό καθεστώς, όπου έχουν υποχρεωτικές και μη υποχρεωτικές δαπάνες, όπου το Συμβούλιο δεν έχει λόγο για τη γεωργία και άλλες υποχρεωτικές δαπάνες, αλλά μόνο τον τελευταίο λόγο για τις μη υποχρεωτικές ε, δαπάνες. Φαίνεται σαν το Συμβούλιο να εξακολουθεί να ζει σε εκείνο τον κόσμο, που το μόνο που πρέπει κανείς να συμφωνήσει είναι κάποια λίγα σημεία και μετά το Κοινοβούλιο μπορεί να ακολουθήσει τα υπόλοιπα. Η ιδέα με την συνθήκη της Λισαβόνας θα έπρεπε να είναι ότι είμαστε επίσης όρις και ότι θα πρέπει να διαπραγματευτούμε αν σειρά προς σειρά, γραμμή προς γραμμή, μέχρι όλες τις λεπτομέρειες, να πούμε τι είναι σοβαρό και τι στέκει και τι όχι. Και αυτό που θα προσπαθήσουμε να κάνουμε αυτή τη φορά είναι λοιπόν να αναγκάσουμε την Ιρλανδική και την Λιθουανική Προεδρία να ακολουθήσουν μια σωστή διαδικασία. Σε τρεις διαπραγματεύσεις ε, δεν μπορέσαμε να έχουμε συμφωνία τουλάχιστον 12 γιατί είδαμε αυτή την κατάσταση. Το Συμβούλιο δεν ήταν έτοιμο να διαπραγματευτεί μέχρι την τελευταία στιγμή με αυτές τις 21 μέρες που είναι η προθεσμία για να πάει κανείς σε διαπραγματεύσεις και έπειτα δεν μπήκε σε λεπτομέρειες. Οπότε πρέπει να γίνουν ακόμα πολλά για το πώς ε, θα πρέπει να προχωρήσουμε και πώς θα μπορέσουμε να συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα με σοβαρότητα. Τώρα, για τη δική σας επιτροπή, πέρα από αυτά τα γενικά, τις γενικές παρατηρήσεις, είναι ενδιαφέροντα κάποια προγράμματα για την ηθαγένεια και για την πολιτική στήριξη για τις ε, τα πολιτικά κόμματα αλλά και οι διοικητικές δαπάνες που μπορεί να είναι πολύ ενδιαφέρον θέμα. Γιατί δεν έχουμε λύσει ακόμα το θέμα. Το Κοινοβούλιο επανειλημμένως έχει ζητήσει από την Επιτροπή και από το Συμβούλιο τι αποφάσισε τελικά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αλλά δεν έχουμε λάβει συγκεκριμένα στοιχεία. Ίσως λοιπόν να έχουμε πολύ σφιχτό κορσέ για τις διοικητικές δαπάνες και όλοι το επιθυμούν αυτό βέβαια. Αλλά τελικά πρέπει τα θεσμικά όργανα να μπορούν να λειτουργήσουν. Και αν δεν αποφασίσει κανείς κάποια διαρθωτικά πράγματα, μπορεί να μην ε, ε, βγάζει το μήνα που λέμε. Γι' αυτό για αυτή την Επιτροπή, όπως και για την Επιτροπή Προπολογισμού, σημαντικό θέμα είναι οι διοικητικές δαπάνες. Είναι ρεαλιστικές. Με αυτό τα λόγια θα σας πω ότι ήρθα να σας ακούσω ε, και ότι φυσικά να σας πω ότι θα είμαστε σε διαρκή επαφή καθώς θα προχωράμε στην δημοσιονομική διαδικασία ε, γιατί το Κοινοβούλιο έχει ένα πολύ καλό τρόπο συνεργασία με τι κοινοβουλευτικέ επιτροπέ και την Επιτροπή Προπολογισμού, πράγμα που σημαίνει ότι είμαστε προετοιμασμένοι και εξοπλισμένοι για διαπραγματεύσει ανά γραμμή του προπολογισμού. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και τώρα θα δώσω το λόγο στον συνάδελφο Μέσερ Σμιτ. Ευχαριστώ κυρία Γέντσεν. σας ευχαριστώ που ήρθατε, που μας παρουσιάσατε και τις προτεραιότητες αλλά και τις διαδικασίες. Είμαστε πολύ ευγνώμονες και είναι πολύ χρήσιμα όλα αυτά. Όσον αφορά για το 2014, όντως πρόκειται για ένα έτος ε, εκλογών. Τα κονδύλια εδώ είναι περιορισμένα και είναι πολύ σημαντικό να συζητήσουμε και να θέσουμε ορθά τις προτεραιότητες ποιες είναι οι σημαντικές μας προτεραιότητες. Σίγουρα θα υπογραμμίσω τρεις ή τέσσερις. Πρώτον, ξεκινάμε την πρωτοβουλία για τους Ευρωπαίους πολίτες, την πρωτοβουλία των Ευρωπαίων πολιτών. Και φυσικά πρόκειται για ένα πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο στα πλαίσια των ε, δημοκρατικών δυνατοτήτων που μας δίνει η νέα συνθήκη. Είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε ποιες είναι οι δυνατότητες, ποιες είναι οι νέες δυνατότητες όσον αφορά το επιχειρησιακό κομμάτι, παραδείγματος χάρη, ποιες είναι οι δυνατότητες αυτού του εργαλείου, τι παραπάνω μπορούμε να κάνουμε. Και βεβαίως όλα αυτά θα πρέπει να ξεκαθαριστούν στην τελική συμφωνία. Δεύτερον, τα πολιτικά κόμματα. Είναι ένα θέμα το οποίο συνεχίζεται συνεχίζουμε συγγνώμη να το επεξεργαζόμαστε, να το συζητούμε και, και για μένα αλλά και για τους περισσότερους μέλη εδώ της Επιτροπής μας πρέπει να βρεθεί μια λύση που να λαμβάνει υπόψη της την αρχή της αναλογικότητας, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων. Θα πρέπει να καταπολεμήσουμε κάθε είδους διακρίσεις και αυτό θα φανεί και από τις προτεραιότητες που θα θέσω στην πρώτη μου γνωμοδότηση. Επίσης, μια άλλη πολύ σημαντική προτεραιότητα είναι η αξιολόγηση που πρέπει να γίνει. Κάθε τόσο γίνεται μια αξιολόγηση. Το 2014 θα πρέπει να επανέλθουμε στο θέμα της ε, συνεισφοράς των ε, πολιτών μας και θα πρέπει να δούμε αυτές οι πρωτοβουλίες πώς έχουν ε, μέχρι τώρα αποφέρει κάποια ωφέλη στους Ευρωπαίους πολίτες, τι έχει αξιολογηθεί θετικά και πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση το 2014. Τέλος, τελευταία πρωτοβουλία, συμφωνώ απολύτως όσον αφορά το διοικητικό κόστος. Βεβαίως, και εδώ νομίζω θα συμφωνήσουν οι περισσότερες πολιτικές ομάδες γιατί στις συζητήσεις που έχουμε μεταξύ των ε, συντονιστών αλλά και των σκιωδών εισηγητών έχουμε μία κοινή προσέγγιση. Τέλος, τελευταία πρωτοβουλία, τελευταίος τομέας που θα ήθελα να προσέξουμε είναι ότι πραγματικά όταν συζητούμε την ε, διαδικασία του προϋπολογισμού θα πρέπει να είμαστε διαφανείς, θα πρέπει να δείξουμε μια ανοιχτή διαδικασία, ιδιαίτερα όταν συζητάμε τις δαπάνες μας, ε, τα έξοδα για τις μετακινήσεις μας, γιατί πρόκειται για χρήματα του Ευρωπαίου φορολογούμενου και είναι πάρα πολύ σημαντικό να είμαστε ανοιχτοί και διαφανείς ως προς αυτές τις δαπάνες. Βεβαίως, επαναλαμβάνω, εδώ μιλώ εξ ονόματός μου, εκφράζω τη δική μου άποψη. Θα πρέπει να συζητηθεί με όλους τους συναδέλφους από τις άλλες πολιτικές ομάδες, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα συμφωνήσουμε και πριν το Μάιο, πριν την προθεσμία που μας θέσατε, θα είμαστε σε θέση να θέσουμε την κοινή μας άποψη. Ο κύριος Νταφ, πρόεδρε. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το Κοινοβούλιο να εκφράσει τις απόψεις του φέτος, καθότι δεν το μπορέσαμε, δεν το καταφέραμε πέρσι. Σήμερα έχουμε την συνθήκη της Λισαβόνας, η οποία έχει τεθεί σε ισχύ και οι διαδικασίες έχουν ε, πλέον προχωρήσει όσον αφορά τον ε, καθορισμό του ετήσιου προϋπολογισμού. Η Ιρλανδική Προεδρία μπορεί σήμερα να προχωρήσει και αυτό καθότι έχει και την ε, ενισχυμένη θέση που προκύπτει από την διοργάνωση δημοψηφισμάτων. Αυτό βεβαίως σήμερα μας οδηγεί στην συνειδητοποίηση των δικαιωμάτων του Κοινοβουλίου όσον αφορά τη διαδικασία του προϋπολογισμού και την δυνατότητα προσφυγής στο δικαστήριο. Υπάρχει ένα προηγούμενο και είμαι σίγουρος ότι το δικαστήριο θα μας στηρίξει. Και αν υπάρξει παραβίαση της συνθήκης, θα ενισχυθεί η δική μας θέση και όχι αυτή του Συμβουλίου. Τώρα, ως προς την ουσία, όπως είπε ο κύριος Μέσερ Σμιτ, πρόκειται για ένα καθοριστικό έτος για όλους μας. Πρόκειται για ένα έτος εκλογών. Άρα όλη η περίοδος που θα οδηγήσει στις εκλογές θα έχει σαν συνέπεια κάποια αυξημένη δραστηριότητα. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε σε θέση να πετύχουμε σε σημαντική προσέλευση στις ευρωπαϊκές εκλογές, δεν θα πρέπει να αυξηθεί ακόμα περισσότερο η αποχή, πρόκειται για θέμα αξιοπιστίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να στοχεύσουμε σε μια προεκλογική εκστρατεία η οποία να κινητοποιήσει τους Ευρωπαίους εκλογές. Δεν έχουν σηκώσει άλλοι το χέρι τους. Πάρα πολύ σύντομα. Γιατί βεβαίως δεν αποφασίζουμε αυτή τη στιγμή τίποτα το συγκεκριμένο και είμαστε στα πρώτα στάδια ε, της συζήτησης και γιατί βεβαίως δεν αποφασίζουμε για σημαντικά θέματα εμείς εδώ σε αυτήν την Επιτροπή. Αλλού λαμβάνονται σημαντικές αποφάσεις ε, με σημαντικές επιπτώσεις στο προϋπολογισμό. Όπως είπε όμως ο κύριος Μέσσερσμιτ, και εμείς ε, ενδιαφερόμαστε να μπορούμε να αποδείξουμε ότι κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να είμαστε προσεκτικοί όσον αφορά τις δαπάνες. Χρειάζεται λοιπόν διαφάνεια, χρειάζεται προσοχή και από την άλλη μεριά η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται κάποιους πόρους, αυτούς τους πόρους ε, πρέπει να τους έχει. Είναι δύσκολο αυτό να πετύχουμε αυτήν την ε, ισορροπία, αλλά είμαι πεπισμένος και ελπίζω ε, με την καλή θέληση που μας χαρακτηρίζει όλους να το πετύχουμε. Έχουμε πάντως μια πολύ σημαντική ευθύνη και θα πρέπει πραγματικά να αξιολογήσουμε όλες τις προσπάθειες που έχουν γίνει μέχρι τώρα, η πρωτοβουλία των πολιτών, το θέμα της ευρωπαϊκής ε, κότητας. Όπως ανέφερε ο κύριος Μέστερσμιτ, η αξιολόγηση αυτών των πρωτοβουλίων είναι πάρα πολύ σημαντική. Επίσης, η επικοινωνία οι κατευθυντήριες γραμμές για την ε, επικοινωνία και την πληροφόρηση. Πολλές φορές η επικοινωνία δεν στοχεύει σωστά. Νομίζω λοιπόν ότι θα αποφασίσουμε καλύτερα και πιο ορθά αν μπορέσουμε να βασιστούμε σε κάποια απτά αποτελέσματα αξιολογήσεων. Γιατί και σαν Κοινοβούλιο και σαν ε, Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αυξήσουμε στο μέλλον τους ίδιους πόρους μας, οι οποίοι θα προέρχονται, όπως πολύ σωστά ακούσαμε, από τον Ευρωπαίο Φορολογούμενο. Και για να γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει πραγματικά να δείξουμε την ικανότητά μας να είμαστε προσεκτικοί και να κάνουμε σημαντικές εξοικονομήσεις. Ένας από τους συνεργάτες μου μου έδωσε κάποια στοιχεία επιπλέον, <clears throat> αλλά δεν ε, λέει τις πηγές αλλά εδώ διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση που δεν συμφωνήσει με τη νέα πρόταση του MFF το Κοινοβούλιο, τότε θα πρέπει η Επιτροπή να κάνει πρόταση για τον προϋπολογισμό του 2014 και η εφαρμογή των ανωτάτων ορίων που ισχύαν τον προηγούμενο χρόνο θα ισχύσουν και για το 2014. Αυτό σημαίνει μια παράταση ουσιαστικά των ορίων του 2013 προσαρμοσμένων με ένα αποπληθωριστικό δίκτυ 2%. Δεν ξέρω τι είδους μεταφράσεις από και προς την Αλβανική έχουν μεσολαβήσει, αλλά καταλαβαίνετε ό,τι καταλαβαίνω και εγώ. Πριν δώσω το λόγο στην κυρία Γένσεν θα ήθελα να πω ότι είναι σωστό αυτό που είπε ο κύριος Νταφ. Υπέγραψε τη μεγάλη σημασία, καθοριστική σημασία που έχει για την περαιτέρω πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης των επομένων εκλογών. οι προεκλογικές εκστρατείε που δεν θα γίνουν μόνο από τα μεμονωμένα κόμματα αλλά και από το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να οδηγήσουν τον κόσμο να ψηφίσει. Και για να το πετύχουμε αυτό πρέπει να δούμε ακριβώς πόσες, ε, τι, τι ποσά απαιτούνται Ήδη τον Μάιο θα πρέπει να δείξουμε τη μεγάλη σημασία που έχει η Ευρώπη και τη μεγάλη σημασία που έχει η συμμετοχή των Ευρωπαίων ε, στις εκλογικές διαδικασίες. Για την πρωτοβουλία των πολιτών, εδώ αναφέρθηκε σε αυτό συγκεκριμένα ο κύριος Μέσερ Σμιτ. Στα πλαίσια της πρώτης εμπειρίας την οποία έχουμε, οι οργανωτές αυτών των πρωτοβουλειών αντιμετώπισαν δυσκολίες για τη λειτουργία του, του συστήματος πληροφορικής. Το σύστημα έτσι όπως προβλέπετε δεν λειτουργεί σωστά. Εγώ δεν τα πολύ καταλαβαίνω αυτά λέει ο Πρόεδρος, αλλά παρόλα αυτά υπάρχει ένα σύστημα το οποίο δίδει τις εγγυήσεις οι οποίες απαιτούνται έτσι ώστε να μην υπάρχουν επαναλήψεις ψήφων κτλ. Αυτό είναι κάτι το οποίο κοστίζει βέβαια στις οργανώσεις των πρωτοβουλειών αυτών και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει ένα σύστημα το οποίο να μπορούν να χρησιμοποιούν έγκυρα και έγκαιρα βέβαια οι οργανωτές των πρωτοβουλειών. Το σύστημα αυτό είναι προσωρινό, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα διατηρηθεί και στο μέλλον. Ε, θα πρέπει να δούμε ακριβώς τι θα γίνει, εν πάση περιπτώσει, με αυτό το σύστημα, έτσι ώστε το σύστημα αυτό της τηλεσυμμετοχής, αν θέλετε, να είναι εύκολο, αξιόπιστο και διαρκές, χωρίς να αυξάνει συνεχώς το κόστος. Νομίζω ότι αυτό δεν είναι κάτι το τρομερά δύσκολο, πρέπει όμως να το υπογραμμίσουμε. Α, κοιτάξτε, έχει ζητήσει το λόγο πάλι ο κύριος Έφνα. Ευχαριστώ. Δύο παρατηρήσεις θα ήθελα ακόμα να κάνω, συμπληρωματικά, οι οποίες έχουν σχέση μεταξύ τους. Έχω την εντύπωση ότι κάποιες φορές, όταν αναφερόμαστε στο προϋπολογισμό για την επικοινωνία, θέτουμε λανθασμένες προτεραιότητες. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Παλιότερα είχα προτείνει να μιλήσουμε για την πρωτοβουλία των Ευρωπαίων ε, πολιτών και να οργανώσουμε μία εκστρατεία που να εξηγεί στους πολίτες της Ευρώπης λέγοντάς τους ότι πραγματικά αυτό που μας ενδιαφέρει είναι οι ιδέες τους για την Ευρώπη. Προτείνετε μας λοιπόν, δώστε μας τις ιδέες σας για την Ευρώπη. Και αν θέλετε αυτό θα έπρεπε να συμπεριληφθεί σε αυτό το οποίο θέλαμε να κάνουμε σαν ενημερωτική εκστρατεία για την πρωτοβουλία αυτή. Φαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν τον θεώρησε ότι ήταν αρκετά σημαντικό σαν σκοπός. Ο κατόπιν ξεκίνησε μια ενημέρωση, δεν είχε γίνει καμία δοκιμή, καμία προετοιμασία. Δεν καταλαβαίνω γιατί. Και τελικά ελέ, ελάχιστα, αν θέλετε, πράγματα έφτασαν μέχρι εμάς. Και γι' αυτό λίγα πράγματα χρειάζονται, λίγα μέσα, λίγη χρηματοδότηση. Ε, αυτό που θέλουμε είναι να παρατηρήσουν οι Ευρωπαίοι πολίτες ότι υπάρχουμε να προσέξουν ότι ζητάμε την απόψή τους και αυτά τα οποία μας προτείνουν να τα χρησιμοποιήσουμε γιατί τελικά είδαμε ότι μήνες μετά το ξεκίνημα αυτής της πρωτοβουλίας ήταν σχεδόν ανύπαρκτη η αντίδραση από μέρους των πολιτών. Αυτό είναι κρίμα και πολλές φορές για ελάχιστα, αν θέλετε, κονδύλια τα οποία θα μπορούσαν να είχαν χρησιμοποιηθεί, τελικά το αποτέλεσμα ήταν ασήμαντο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πολλές φορές χρησιμοποιεί πολύ σημαντικότερα κονδύλια. Το αποτέλεσμα, επαναλαμβάνω, δεν είναι αυτό που περιμέναμε. Δεν είναι αποτελεσματική η δράση και βλέπουμε ότι θα πρέπει με ένα πολύ ξεκάθαρο τρόπο να οργανωθεί από εδώ και πέρα. Δεν λέω ότι πρέπει καμία σύμβαση να περνάει από την Επιτροπή, αλλά εν πάση περιπτώσει αν κοιτάξω όλα τα μέτρα, όλες τις ε, διαδικασίες που έχουν αποφασιστεί, έχω την εντύπωση ότι είναι πλέον επίγον να αλλάξει ο τρόπος λειτουργίας ε, τέτοιων ε, ενημερωτικών κινήσεων. Και ίσως θα έπρεπε να σταματήσουμε να λέμε στους Ευρωπαίους «Ελάτε, ψηφίστε, πρέπει να τους δείξουμε ότι μας ενδιαφέρει η άποψή τους, ότι μας ενδιαφέρουν οι Ευρωπαίοι ψηφοφόροι. Να κάνουμε κάποιες εκκλήσεις, μια πιο συγκεκριμένη πληροφόρηση και ενημέρωση και νομίζω ότι ο κόσμος πλέον θέλει ουσία. Well, thank you very much. Well, I think the Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω πως ε, η συζήτηση περί της πρωτοβουλίας των πολιτών δείχνει ότι κατά πόσο θα έπρεπε να υπάρχει μια γραμμή του προϋπολογισμού ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια για τους πόρους που θα κατανεμηθούν ακριβώς για αυτό το στόχο. Θα έλεγα λοιπόν να συνεχίσετε σε αυτό το πνεύμα. και πιστεύω πως ίσως αυτό να είναι το βασικό πρόβλημα μαζί με τις εκλογές του χρόνου. Εγώ δεν είμαι η συγκήτρια για τα άλλα θεσμικά όργανα, Συμβούλιο, δικαιο, Δικαστήριο. Είναι η κυρία Χόλμαϊρ. Και η οποία φυσικά θέλει να κάνει ε, οικονομίες και έχει βάλει για αυτό το θέμα ψηλά στην ημερήσια διαταξή. Σε σχέση με αυτό που ανέφερε ο κύριος Πόνς ε, για το ε, αν θα μπορούμε εμείς να δώσουμε τη συγκατάθεσή μας ή όχι, Ας ελπίσουμε ότι μέσω των διαπραγματεύσεων θα βρούμε μια λύση ειρηνική για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, γιατί αν δεν το καταφέρουμε αυτό τότε θα είναι η οροφές του 2013 που θα ισχύσουν για το 1η Ιανουαρίου του 2014. Είναι γεγονός δε ότι για το 2014 δεν είμαστε και πολύ μακριά από τις προτάσεις της Κομισιόν για το PDP. Γίνονται όλο και πιο παράξενο καθώς προχωράμε, γιατί είναι πολλά για τη Γεωργία και πολύ λίγα για τα άλλα κομμάτια του προϋπολογισμού που αφορούν την ανάπτυξη, την έρευνα, την παιδεία, ε, και τις υποδομές. Καθώς λοιπόν περνά ο χρόνος, τόσο χειρότερο είναι για πολλούς από εμά που θα θέλαμε να υπάρξει μεγαλύτερη ε, επικέντρωση στην ανάπτυξη. Μπορούμε να τα καταφέρουμε, αλλά φυσικά είναι καλύτερο να βρούμε μια λύση. Και στις κατευθυντικές γραμμές λέγεται, αναφέρεται, πως η Κομισιόν παίρνει ως βάση την πρόταση που έκανε για το πολιετές δημοσιονομικό πρόγραμμα δεν ήταν πλειοψηφία, δεν ήταν η πλειοψηφία της Επιτροπής Προϋπολογισμού που ήθελε να υπογραμμίσει ότι δεν δεχόμαστε τα αποτελέσματα τα μάλλον τα πορίσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Είμαστε υπό διαπραγματεύσει. Αυτό είναι ίσως το υπόβαθρο για τι διαπραγματεύσει. Αυτή είναι η πρόταση της Κομισιόν και φυσικά αυτό μπορεί και να αλλάξει. Τώρα για τη διαδικασία από εδώ και στο εξή μπορούμε να πούμε ότι μπορεί να υπάρξει μια καθυστέρηση για την πρόταση της Κομισιόν γύρω στα μέσα Μαΐου το αναμένουμε ή τέλος Μαΐου θα δούμε. Ίσως αυτό να μην ε, μας ε, διευκολύνει, να δούμε δηλαδή πώς θα κάνουμε τις αλλαγές. και πώς θα ψηφίσει το Συμβούλιο τον Αύγουστο, γιατί επιμένει να ερμηνεύει τη συνθήκη του, της Λισαβόνας με τέτοιο τρόπο ώστε αν έχει έναν προϋπολογισμό κάθε φορά να πρέπει να το στέλνει σε όλα τα εθνικά κοινοβούλια για να δεις αν πιστεύουν ότι θα πρέπει να έχει Ευρωπαϊκή Ένωση προϋπολογισμό για του χρόνου και πάντοτε το κάνουν αυτό το καλοκαίρι όπου κανείς δεν απαντά. Αλλά είναι παράξενο να έχουμε αυτή την καθυστέρηση. Πάντως, έτσι επέλεξε να τρομινεύσει ε, το Συμβούλιο. Και πάντως προσβλέπουμε στη συνεργασία με την ε, Επιτροπή σας. Ωραία, σας ευχαριστούμε κυρία Γένσεν για αυτή την ε, συνάντηση. Ξέρω, επισκέπτεστε όλες τις επιτροπές. Σας ευχαριστώ και κλείνει αυτό το σημείο στην ημερήσια διάταξη. <laughs> E Περνάμε στο επόμενο σημείο στη μερισσία διάταξη, την έκθεση Γκουερέρο για την τροποποίηση του κανονισμού 967 του 12 σχετικά με τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων. Η Επιτροπή Προϋπολογισμών και η κυρία Γκρέσλε είναι αρμόδια επί της ουσίας. Εμείς θα εκφέρουμε μία γνωμοδότηση σήμερα, την οποία θα την διατυπώσει ο κύριος Γκοερέρο. Κανονικά είχαμε πει ότι θα ψηφίζαμε για την έκθεση Γκορμάη, θα περιμέναμε την έκθεση Γκορμάη, αλλά είναι ήδη σε θέση ο κύριος Γκουερέρο να παρουσιάσει την γνωμοδότησή του. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θεωρώ δεδομένο ότι όλα τα μέλη της Επιτροπής γνωρίζουν επαρκώς τη διασύνδεση ανάμεσα στην έκθεση της κυρίας Γιαννάκου και την τροποποίηση των δημοσιονομικών κανονισμών. Στην ουσία, αλλάζοντας το καθεστώς της χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων, στα πλαίσια και της έκθεσης της κυρίας Γιαννάκου που κανονικά θα ψηφίσουμε αύριο, θα καταστεί απαραίτητο να τροποποιήσουμε και τις ε, οικονομικές ρυθμίσεις, οι δημοσιονομικές ρυθμίσεις που εφαρμόζονται στο τμήμα της εκθέσεως της κυρίας Γιαννάκου που έχει σχέση με τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων. Θα πρέπει να συζητήσουμε θέματα επί της ουσίας. <clears throat> σχετικά με την χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων. Πάνω σε αυτό έχουν εκφραστεί ε, διαφορετικές απόψεις και διαφορετικοί τρόποι αντίληψης, θα έλεγα, του θέματος. Και αυτό είναι μια συνέπεια θα έλεγα μηχανιστικού τύπου της κατάστασης. Απ' τη μία υπάρχουν ορισμένες ρυθμίσεις οι οποίες αφορούν την έκθεση της κυρίας Γιαννάκου και αυτό μπορεί να γίνει μέσω της προσαρμογής των κανόνων, των δημοσιονομικών, κάτι το οποίο έχει άμεση σχέση με την τροποποίηση του καθεστώτος του ιδίου της λειτουργίας των πολιτικών κομμάτων. Ελπίζουμε λοιπόν, θα πρέπει να περιμένουμε μάλλον την έκθεση, την έκθεση της κυρίας Γιαννάκου για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τις ε, οικονομικές, αν θέλετε, την εικόνα για το σύνολο των οικονομικών αλλαγών που θα πρέπει να υπάρξουν. Η Επιτροπή Προϋπολογισμών όμως, η οποία είναι υπεύθυνη επί της ουσίας, έχει ήδη προχωρήσει σε μια προσωρινή έκθεση την οποία δεν θα εγκρίνει επίσημα όσο δεν έχει ολοκληρωθεί η πορεία της εκθέσεως της κυρίας Γιαννάκου. Και έτσι λοιπόν μπορούμε με βάση αυτή την προσωρινή έκθεση και με βάση τις τροπολογίες οι οποίες θα κατατεθούν, μπορούμε να κάνουμε μια πρώτη συζήτηση, γνωρίζοντας όμως ότι δεν θα κάνουμε καμία ψηφοφορία για το θέμα αν δεν ολοκληρωθεί η διαδικασία της εκθέσεως της κυρίας Γιαννάκου. Συνεπώς, αυτό το οποίο έχω ήδη πει, περιλαμβάνει κάποιες γενικές ε, σκέψεις για το πόσο επίκαιρο είναι να υπάρξει ένα ενιαίο καθεστώς για τα κόμματα ευρωπαϊκού μεγέθους αν θέλετε Επίσης να υπάρχει μια χρηματοδότηση αυτών των οργανισμών των πολιτικών έτσι ώστε να αποτρέπονται κάποιες διακρίσεις οι οποίες συνήθως συμβαίνουν στην περίπτωση που υπάρχουν και ιδιωτικές μορφές χρηματοδότησης και ταυτόχρονα υπογραμμίζουμε την ανάγκη που υπάρχει να προσαρμόσουμε στις ε, καθημερινές πολιτικές σχέσεις μας και να ενημερώσουμε σωστά την διαχείριση και τον έλεγχο της οικονομικής αυτής λειτουργία των πολιτικών κομμάτων που θα πρέπει να είναι διαφανέστατη και να ελέγχεται από τους ε, ευρωπαϊκούς οργανισμούς, από τα ευρωπαϊκά όργανα. Πρόκειται λοιπόν σε αυτή τη φάση για ένα έγγραφο εργασίας ουσιαστικά, στα πλαίσια του οποίου εγώ ε, στηρίζω τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τις σχετικές με την αλλαγή του συστήματος ε, των otro sistema más moderno que recibe el nombre de contribuciones να υπάρχουν από τη μία το σύστημα των συνασφορών και από την άλλη το σύστημα των άμεσων επιδοτήσεων. Νομίζω ότι το σύστημα το οποίο λειτουργούσε μέχρι τώρα, σύμφωνα με το οποίο κάθε χρόνο πρέπει να παρουσιάζεται ένα πρόγραμμα εργασίας και έτσι να μπορεί να καλύπτεται η ευελιξία την οποία έχουν ανάγκη τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα. Αυτό θα πρέπει να αλλάξει έτσι ώστε να υπάρχει μια ενιαία παρουσίαση της οικονομικής διαχείρισης των πολιτικών αυτών οργανισμών στο τέλος της περίοδου. Υπήρξαν και άλλες ανταλλαγές απόψεων ε, σαν παράδειγμα τι θα γίνει με τα υπόλοιπα τα οποία δεν έχουν δαπανηθεί κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης χρονικής περίοδου από ορισμένα πολιτικά κόμματα. Θα δίδεται μια προθεσμία διετή σαν παράδειγμα στους πολιτικούς αυτούς τους οργανισμούς έτσι ώστε να τεκμηριώνουν τη χρήση ημί των συγκεκριμένων ποσών. Λοιπόν είμαι επίσης υπέρ του να μειωθεί το ποσοστό συγχρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων, έτσι ώστε για να αποφύγουμε για μια ακόμη φορά τα κόμματα τα οποία λαμβάνουν μικρότερες ιδιωτικού τύπου χρηματοδοτήσεις, ιδιωτικού τύπου επαναλαμβάνω, να μην βρίσκονται σε χειρότερες καταστάσεις και να αντιμετωπίζουν περισσότερες δυσκολίες από ότι τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα. Παρατηρώντας τώρα τις τροπολογίες θα δείτε ότι υπάρχει μια συνεχής μόνιμη αναφορά σε μια απόφαση, ε, σε μια έκθεση καλύτερα του ελεγκτικού συνεδρίου που ε, χρησιμεύσε στην Επιτροπή προϋπολογισμών έτσι ώστε να επεξεργαστεί την δική της έκθεση, την πραγματική κοινοβουλευτική της έκθεση, ενώ εμείς επαναλαμβάνω εδώ δεν κάνουμε παρά μία γνωμοδότηση. Εγώ θα ήθελα να πω ότι συμπίπτω εν πολλής με τις προτάσεις της Επιτροπής ε, Προϋπολογισμών και με τη σειρά της η Επιτροπή Προϋπολογισμών συμπίπτει εν πολλής ε, με τις αποφάσεις τις οποίες κατέληξε το ελεγκτικό συνέδριο. Σύμφωνα με τις αποφάσεις αυτές δεν θα πρέπει να υπάρξει μια ιδεολογική συζήτηση, το θέμα είναι πρακτικό θα πρέπει να δούμε με βάση την εμπειρία που έχει το ελεγκτικό συνέδριο το πώς θα ελέγξουμε καλύτερα την χρηματοδότηση και κάθε μορφή και τρόπο χρηματοδότησης των πολιτικών ευρωπαϊκών κομμάτων με τα οποία ασχολείται με άλλο τρόπο όμως η κυρία Γιαννάκο. Λοιπόν, υπάρχει κάποιος χρόνος, κάποια διαθεσιμότητα και από πλευράς μου για να συζητήσουμε τις τροπολογίες τις οποίες θα μου αποστείλουν στο μέλλον τα μέλη της Επιτροπής μας. Να αναφερθώ στο χρονοδιάγραμμα. Το χρονοδιάγραμμα έτσι όπως προβλέπετε τώρα είναι σήμερα να κάνουμε την παρούσα συζήτηση η οποία είναι μια προκαταρκτική συζήτηση θα υπάρξει μια προθεσμία για την κατάθεση των τροπολογιών από πλευρά των ε, συντονιστών που κανονικά δεν θα πρέπει να ξεπεράσει την 22η Απριλίου. για να έχουμε τη δυνατότητα να τη συζητήσουμε άπαξ και την επομένη 23 Απριλίου να μπορέσουμε να ψηφίσουμε έτσι ώστε να συμπέσουμε χρονικά και με την έγκριση από πλευράς της Επιτροπής Προϋπολογισμών της εκθέσεώς της, της κύριας εκθέσεώς της, η οποία προβλέπεται για τις 26 Απριλίου. Έχουμε λοιπόν κάποιο χρόνο μέχρι τις 22 Απριλίου για την κατάθεση των τροπολογιών. Έχουμε χρόνο για να προσπαθήσουμε να πετύχουμε κάποιους συμβιβασμούς όπου αυτό χρειάζεται. 22 του μηνός θα τεθεί το θέμα στην ΑΦΚΟ επίσης Εγώ δεν ξέρω αν πιστεύετε ότι ε, είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξο πάνω σε αυτό. Έχω όμως παρόλα αυτά την αίσθηση ότι δεν θα πρέπει να δημιουργηθούν πάρα πολύ ε, δύσκολες καταστάσεις με στα πλαίσια της συζήτησης της νομοδότησης αυτής. Η ουσία του πράγματος βρίσκεται στην έκθεση της κυρίας Γιαννάκου και στη συγκεκριμένη περίπτωση, στην περίπτωση της νομοδοτήσεώς μου, τίθεται περισσότερο το θέμα με λογιστικό θα έλεγα τρόπο. Είναι θέμα πρακτικό και είναι κάτι το οποίο συνδέεται με την μεγάλη εμπειρία την οποία έχει το ελεγκτικό συνέδριο γύρω από τα θέματα αυτά. Προτείνω λοιπόν και με τις τοπολογίες όχι μόνο να συνεργαζόμαστε στενά με το ελεγκτικό συνέδριο, αλλά επίσης να συνεργαζόμαστε στενά και με την ΟΛΑΦ, να προσπαθούμε να είμαστε όσο περισσότερο ευέλικτοι γίνεται και να διασφαλίσουμε έτσι έναν αυστηρότατο έλεγχο των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων. Ο κύριος Ντάφ έχει ζητήσει το λόγο. Πρόεδρε να ευχαριστήσω για τις ε, εξηγήσει ε, και συμφωνώ τόσο ότι πρέπει πραγματικά να παρακολουθήσουμε το θέμα και να ακούσουμε τις προτάσεις ε, του ελεγκτικού συνεδρίου. Όντως ε, η αναβολή της ε, ψηφοφορίας ε, για την έκθεση Γιαννάκου έτσι κι αλλιώς είχε προταθεί και αποφασιστεί γιατί όπως είπαμε δεν είχαμε την εντύπωση ότι το θέμα είχε οριμάσει αρκετά, ότι η συζήτηση είχε ολοκληρωθεί και αυτό δυσκολεύει βέβαια κατά κάποιο τρόπο την απόφαση και το χρονοδιάγραμμα. Θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση. Για ποιο τμήμα του Κοινοβουλίου νομίζετε ότι θα πρέπει να παίξει το ρόλο της αρμόδιας αρχής όσον αφορά την, τις συνεισφορές αυτές. Στην πρότασή σας βλέπω ότι υπάρχει μια σχετική διακριτική ευχέρεια και ότι κάποιος θα είναι αυτός ο οποίος θα αποφασίζει Πώς πιστεύετε εσείς ότι πρέπει να οργανωθεί το Κοινοβούλιο έτσι ώστε να εφαρμοστούν αυτοί οι κανόνες. Δεύτερη ερώτηση. Πιστεύετε ότι θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα μίας διαδικασίας προσφυγής σε περίπτωση, παραδείγματος χάρη, που ένα από τα εμπλεκόμενα μέρη θεωρεί, παραδείγματος χάρη, ότι δεν έχει υποστηριχθεί ιδεόντως ή ότι του έχουν στηριχθεί κάποια από τα κονδύλια που θα έπρεπε να είχε πάρει. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια τέτοια δυνατότητα προσφυγής ή δεύτερης εξέτασης. Μπορούμε να σκεφτούμε κάποια τέτοια διαδικασία. Δεν έχω να ζητήσει άλλη το λόγο και γι' αυτό θα δώσω στον κύριο Γκουερέρο τη δυνατότητα να απαντήσει. Να πω επίσης και προς τον κύριο Νταφ Υπάρχει ένα θέμα σχετικά γενικό εδώ. Μιλάμε για τον λεγόμενο authorizing officer, τον διατάκτη, αλλά δεν εξηγούμε περί ποιου πρόκειται. Η γενική ιδέα την οποία έχουμε είναι να προσπαθήσουμε να μην περιπλέξουμε τα πράγματα περισσότερο. Οπότε κανονικά η ίδια η Γενική Γραμματεία του Κοινοβουλίου είναι αυτή, η οποία θα κληθεί να δώσει απαντήσεις και σε σχέση με το δεύτερο ερώτημα το οποίο έθεσε ο κύριος Νταφ. Ο μηχανισμός λοιπόν απάντησης θα πρέπει να αναφέρεται κυρίως στη Γενική Γραμματεία του Κοινοβουλίου κάθε φορά. Θα πρέπει όμως, είναι αλήθεια, να διευκρινίσουμε με πιο σωστό τρόπο έτσι ώστε αν η έκθεση για τον προϋπολογισμό δεν περιέχει τις απαιτούμενες διευκρινήσεις, τότε θα πρέπει να προσπαθήσουμε εμείς να επεξεργαστούμε καλύτερα τα πράγματα έτσι όπως το προτείνει ο κύριος Νταφ. Κοιτάξτε λέει ο Πρόεδρος, εδώ μπορούμε να κλείσουμε. Νομίζω ότι μπορούμε να κλείσουμε επίσης και τα διαδικαστικά στα οποία αναφέρθηκε ο κύριος Γκουερέρο. Προθεσμία κατάθεσης των τροπολογιών είναι η 8η Απριλίου 12η Μεσημβρινή, εφόσον συμφωνείτε. Περνάμε λοιπόν τώρα, όπως είπα στην αρχή, ότι έχει αφαιρεθεί από την ημερήσια διάταξη η ευμηνία των άρθρων 156 και 161 του κανονισμού, γιατί δεν έχουν προπαρασκευαστεί σωστά τα έγγραφα τα οποία θα πρέπει να μας απασχολήσουν. Περνάμε στο 7 τώρα. Το 7 αφορά το θέμα της διερμηνίας του 159 του κανονισμού και τι συμβαίνει στην περίπτωση ε, ισοψηφίας. Είχαμε αναφερθεί και στο θέμα της τσεχικής δημοκρατίας και στην αίτηση που είχε τεθεί για την εξαίρεσή της εδώ τίθεται όμως μια συγκεκριμένη ερώτηση από πλευράς της νομικής επιτροπής, η οποία ζητά στα πλαίσια της διαδικασίας της προβλεπομένης από το 128 σχετικά με την παρέμβαση του Κοινοβουλίου στις ε, διαδικασίες ε, ε, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Τι συμβαίνει στην περίπτωση της ψηφοφορίας επί της προτάσεως του εισηγητή να μην παρέμβουμε αν υπάρξει μια πλειοψηφία. Η πλειοψηφία αυτή ε, ε, τι είδους θα πρέπει να είναι. Ζητήσαμε τη γνώμη της νομικής επιτροπής η οποία απαντά ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί το γενικό καθεστώς ψηφοφοριών το προβλεπόμενο από το 159. Δεν προβλέπεται από τον κανονισμό στη συγκεκριμένη περίπτωση καμία απόκληση. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει στη συγκεκριμένη περίπτωση καμία σύσταση από πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν έχω να κάνω κάποιο σχόλιο πάνω σε αυτή τη γνωμοδότηση. Αν η πρόταση του εισηγητή είναι να μην προχωρήσουμε σε δικαστικά μέσα, τότε από εκεί και πέρα δεν υπάρχει απλά καμία δυνατότητα προσφυγής νομικά. Λοιπόν, αυτή είναι η απάντηση το άρθρο 159 παράγραφος 3 του κανονισμού θα πρέπει να ερμηνευθεί με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε στην περίπτωση ισότητας ψήφων κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας εξέτασης μια συστάσεως επί τη βάση του άρθρου 128 παράγραφος 4 περί μη παρέμβασης και συμμετοχή σε διαδικασία προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δεν σημαίνει την υιοθέτηση μιας συγκεκριμένης συστάσεως. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν δεν θα υπάρξει συνέχεια. Νομίζω ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με μια ερμηνεία του πνεύματος και του γράμματος του κανονισμού. Δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα. Η γνώμη μας είναι συμβατή με τη γνώμη της νομικής υπηρεσίας. Νομίζω ότι αν κάποιος θέλει το λόγο Ούτε καν ο κύριος δεν θέλει να πάρει το λόγο στη συγκεκριμένη περίπτωση. Εφόσον δεν υπάρχουν λοιπόν άλλα θέματα, τότε θα θέσουμε την πρόταση αυτή σε ψηφοφορία αύριο κατά τη διάρκεια των προβλεπομένων ψηφοφοριών. Λοιπόν, με αναβολές και αναβολές, για μεγάλη χαρά ορισμένων που χαμογελούν ιδιαίτερα, βλέπω να έχουμε τελειώσει εδώ. Να σας υπενθυμίσω πάντως ότι αύριο στις 9 ε, με 10 έχουμε τη συνάντηση των συντονιστών. Ξέρετε ότι δεν θα έχουμε την ψηφοφορία της εκθέσεως της κυρίας Γιαννάκου. Θα συζητήσουμε κατά τη διάρκεια των συντονιστών τι θα κάνουμε με την πιθανή συζήτηση της εκθέσεως της κυρίας Γιαννάκου. Απλά δεν θα υπάρξει ψηφοφορία. Αυτό θα το αποφασίσουν αύριο λοιπόν οι συντονιστές. Τέλος της συνεδριάσεως. Μπράβο.